και η έκθεση αυτή ενισχύει αυτή τη διάθεσή μας. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Έχει κλείσει η συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα είναι αύριο στις 11 και 30 στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε τώρα την προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν για την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητος μετά τη θέση σε εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Κύριε Σεύκοβιτ, γεια σας. Mm. Δεν με ακούτε, δεν πειράζει. Και δίνω το λόγο στην κυρία Κοχμερίν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, πρόκειται για ένα ερώτημα το οποίο είναι πράγματι επίκαιρο και σημαντικό. Γνωρίζουμε ότι πριν από την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας υπήρχε και το γεγονός ότι 80% αυτών που αποφάσισαν τα εθνικά κοινοβούλια αποφασιζόντουσαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό δεν έχει αλλάξει μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τα, τα εθνικά κοινοβούλια όμως τώρα έχουν ένα σημαντικό ρόλο τον οποίο μπορούν να επομιστούν μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των πολιτών. Και αυτό είναι ενδιαφέρον και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τα εθνικά κοινοβούλια. Αλλά παρόλα αυτά υπήρξαν προσφυγές από τα εθνικά κοινοβούλια γιατί θεωρούν ότι αυξήθηκε ο φόρτος εργασίας τους. Έχουν όλο και περισσότερα έγγραφα τα οποία έρχονται στην, ε, στο τραπέζι τους πρέπει να αντιδράσουν μονάχα σε μερικές εβδομάδες σε όλα αυτά τα νομοθετήματα και η εντύπωση είναι ότι όλο και περισσότερο ζητούνται από τα κράτη-μέλη να εργαστούν περισσότερο. Το απαραίτητο είναι να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει δυνατότητα να αντιδρούν όμως στις πρωτοβουλίες των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν. Μετά λοιπόν από τη θέση εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι όπως και εγώ που θεωρήσαμε ότι αυτό είναι το κατάλληλο χρονικό σημείο για να δούμε πώς ακτιμά την κατάσταση η Κομισιόν αυτή τη στιγμή, κατά πόσο είναι ικανοποιημένη με τις αντιδράσεις που προέρχονται από τα ευρωπαϊκά εθνικά κοινοβούλια, αν θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκή πόρη και επαρκέ προσωπικό στα Εθνικά Κοινοβούλια για να αντιμετωπίσουν την πρόσθετη αυτή εργασία και επίση στην περίπτωση περιφερειακών κοινοβουλίων όπω είναι τα Ομοσπονδιακά κρατήρια στην Γερμανία, αν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με επαρκή τρόπο αυτά τα νέα καθήκοντα και αν υπάρχει μια επαρκή ανταπόκριση από τη δική του πλευρά σε σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο έδωσα μαζί με τον Άντριου Ντάφ και πολλού άλλου συναδέλφου και περιμένω αδειμόνω την απάντησή σα. Ευχαριστούμε κυρία Κόχμερη. Ο κύριο Σεύκοβιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ την αξιότιμη κυρία Βουλευτή για τι ερωτήσει που υπέβαλε. Διότι έτσι μα δίνεται η ευκαιρία να υποβάλουμε την γενική μα εκτίμηση όσον αφορά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου υπαρχμών 2 του προσυρτημένου στην συνθήκη τη Λισαβόνα αλλά και τον επικορικό μηχανισμό ελέγχου. Διότι αυτό ο μηχανισμό ήδη έχει τεθεί ει λειτουργία, η δε εφαρμογή του μέχρι σήμερα ε, πάει πάρα πολύ καλά και αυτό ε, λόγω τη ε, άρτιας προ, από τα κοινοβούλια, από την Επιτροπή πριν τη θέση συνθήκη. Αλλά επίση αυτό οφείλεται και στην άρρητη συνεργασία και τι εκτεταμένε επαφέ μεταξύ Επιτροπή και Εθνικών Κοινοβουλίων. Μέχρι σήμερα η εμπειρία μα έχει καταδείξει ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι όριμα να λάβουν αυτόν τον νέο ρόλο και τι νέε αρμοδιότητε που του απονέμει κυρία Συνήκη. Και κατά τα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει ότι έχουμε 100 39 σχέδια νομοθετημάτων δυνάμει αυτού του μηχανισμού επικουρικού ελέγχου και προς τα Εθνικά Κοινοβούλια και έλαβε 61 αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις και βέβαια είχαμε κάποια τέτοια σχέδια νομοθετημάτων που αντέβαιναν στην επικουρικότητα. Τώρα είχαμε το πρωτόκολλο 2, το οποίο όριζε το πώς θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία της πορτοκαλί κάρτα και δεν θα πρέπει να περιοριζόμεθα ει θέματα επικουρικότητα σχετικά με τον μηχανισμό αυτό. Όμω είχαμε πει εμεί ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε τον πολιτικό διάλογο με τα κοινοβούλια ε, διότι ε, ο διάλογο ε, για σαν μέσο πολιτικής είναι μόνο μία εναλλακτική αυτό ο μηχανισμό. Θα πρέπει επομένω τώρα να δούμε ότι έχουν πάνω από 600 γνωμοδοτήσεις ετησίου από τα Εθνικά Κοινοβούλια και τις γνωμοδοτήσεις που αφορούν το περιεχόμενο της, των δικών μας προτάσεων. Στη Γενική μας Γραμματεία έχουμε ένα τμήμα του προσωπικού που ασχολείται με τις επαφές με τα κοινοβούλια, αλλά και σε κάθε Γενική Διεύθυνση έχουμε συντονιστάς. Αυτή έχουν συμπαθεί με τα Εθνικά Κοινοβούλια και έτσι μπορούμε να έχουμε εύρυθμη εφαρμογή αυτού του μηχανισμού και τη λειτουργία του. Επίσης και στα ιδιαίτερα γραφεία των επιτρόπων υπάρχουν υπάρχει που ασχολούνται με αυτό και θα μπορώ να σας πω ε, εφόλες της ύλης ότι ο πολιτικός διάλογος, ο μηχανισμός ελέγχου στην ΚΟΖΑΚ συζητείται παγίως και συνεχώς. Εκεί προσέρχονται εθνικοί βουλευτές και είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Κύριε Βουλευτή, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να ασχολούνται περισσότερο οι εθνικοί βουλευτέ με αυτέ τι συζητήσει που αφορούν την κοινωτική νομοθεσία. Και επίση διαπιστώθηκε ότι αυτή η προβληματική τελικά ε, οδήγησε σε ποιοτικέ γνωμοδοτήσει των εθνικών κοινοβουλίων. Εμεί θέλουμε να μιμηθούμε τα εθνικά κοινοβούλια στα όσα ασχολούμαστε εμεί, διότι Πολλά από αυτά που ετέθησαν στην Κόζακ αφορούσαν τα σχόλια των κοινοβουλίων και σε μερικά σημεία μας είπαν ότι θέλουν να είμαστε πιο ακριβείς και να εξηγούμε περισσότερο τις ρήτρες επικουρικότητας ή στι δικές μας νομοθετικές προτάσεις και επομένως μαθαίνουν και οι μεν και οι δε. Στην επόμενη φάση θα πρέπει να διαπιστώσουμε κατά πόσον ανατομέα οι προτάσεις που υποβάλλονται, μεταφορές, περιβάλλον κλπ. κατά πόσον θα συζητούνται όχι μόνο στις Ευρωπαϊκέ επιτροπέ, αλλά και στι καθήλυνα αρμόδιε των εθνικών κοινοβουλίων διότι έτσι νομίζουμε ότι θα αναζωοποιηθεί το εθνικό ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή νομοθεσία και επίση έτσι θα είναι τα κράτη-μέλη πιο προσεκτικά με την μεταφορά εις το εσωτερικό δίκαιο του κοινωτικού δικαίου άρα νομίζω ότι ο μηχανισμός θα πάει μια χαρά ο δε πολιτικό Διάλογο είναι πάρα πολύ σοβαρό, μα δίνει τη ευκαιρία να έχουμε τις γνωμοδοτήσεις που θέλουμε, τις ιτιολογημένες και φυσικά έχουμε και feedback, ενθάρρυνση και λοιπά από τα Εθνικά Κοινοβούλια και είμαι βέβαιος ότι και από τις δύο πλευρές και από εμά και από τα Κοινοβούλια θα έχουμε όλο ένα καλύτερες επιδόσεις ή στο άμεσο μέλλον και σας ευχαριστώ. Και εσύ κυρία Φλασίκο μπαίνουμε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, μέσα στα πλαίσια των διαμεμοιρασμένων αρμοδιοτήτων η αρχή της επικορικότητας είναι αυτή που διέπει το πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εκπροσωπήσει την άποψη των κρατών μελών. Η αρχή της επικορικότητας από τη μία πλευρά σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει προστασία των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Συγχρόνως όμως δίδει τη δυνατότητα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει εάν τα κράτη-μέλη δεν κινούνται όταν αδρανούν. Η... Τα εθνικά κοινοβούλια μετά από την θέση σε εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας και ιδίω του πρωτοκόλου 2, αυτό είναι και το αντικείμενο της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση αυτή αντιμετωπίζει τον τρόπο με τον οποίο η αρχή της επικουρικότητας εφαρμόζεται στην πράξη σε ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως είναι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή των Περιφερειών και αναφέρεται επίσης στο ερώτημα του πώς τα εθνικά κοινοβούλια αντιμετωπίζουν και εφαρμόζουν την αρχή της επικουρικότητας μετά την θέση εφαρμογή τη Συνδικής Λισαβόνα. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα πλέγμα ερωτήσεων που αντιμετωπίζουν ακριβώ την αρχή τη επικουρικότητας. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να διατηρήσει και να υπεραμεινθεί τη αρχή της επικουρικότητας. Τα κράτη-μέλη από το 2009 είχαν τη δυνατότητα να πληροφορήσουν την Κομισιόν <clears throat> στην περίπτωση που κάποια από τα νομοθετήματά τους δεν, ε, δεν συμβάδιζαν με την αρχή της επικουρικότητας. Γι' αυτό έγινε και το ερώτημα του πώς η Κομισιόν αξιολογεί όλη αυτή τη διαδικασία κοινοποίηση και πώς πληροφορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπασέσκου για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζω το ότι συζητάμε ξανά την ε, αρχή της επικουρικότητας μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός ελέγχου έτσι ώστε το άρθρο 5 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης να τηρείται μια ξεκάθαρη κατανομή των αρμοδιοτήτων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο κάνει τα πράγματα απλούστερα δηλαδή απλούστερη τη χρήση της αρχής της επικουρικότητας λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω πως το ΔΕΚ δεν έχει έλεγχο για την εφαρμογή αυτής της ε, αρχής μπορεί μόνο να ανακαλέσει μία νομοθετική πράξη χωρίς να διαπιστώσει το εάν εφαρμόστηκε αυτή η αρχή ή όχι. Οπότε έχουμε εδώ πέρα μια συμπλήρωση δραστηριότητα του ΔΕΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το να οικοδομήσουμε την Ευρώπη σημαίνει να ενσωματώσουμε, να συνενώσουμε Θα ήθελα να ζητήσω τον κύριο Επίτροπο να ακούσει τουλάχιστον αυτά τα οποία έχω να του πω. Αν δεν σας πειράζει κυρία Πρόεδρε, μπορώ να ξαναξεκινήσω. Το να οικοδομήσω την Ευρω... οικοδομήσουμε την Ευρώπη, έλεγα κύριε Επίτροπε, σημαίνει να ενσωματώσουμε και να συνενώσουμε και την ε, ομοσπονδιακή ιδέα, το φεδεραλισμό, αλλά και τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Πρέπει να προχωράει η Ευρώπη από κάτω προς τα πάνω και η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις θεσμικές της σχέσεις με τις περιφερειές της. Αυτό το πρωτόκολλο ήταν ένας, μια ευκαιρία για να προχωρήσουμε και δεν έχει τύχει πλήρου εκμετάλλευση. Οι περιφέρειε τη Ευρώπη βρίσκονται πιο κοντά στου πολίτε και έχουμε πολλά πράγματα να του προσφέρουν. Η Επιτροπή Περιφερειών θεωρεί ότι θα πρέπει τουλάχιστον οι απόψει τη ε, Επιτροπή των Περιφερειών να περιλαμβάνονται στι εκθέσει επικουρικότητα. Σε μία γραπτή απάντηση το Συμβούλιο του προηγούμενου μήνα μου είπε ότι δεν έχει καθόλου πληροφορίε για το πώ τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν τι ανησυχίε των περιφερειών του. Το ίδιο μου και το 2010. Ούτε γνωρίζει το Συμβούλιο ποιε είναι οι θέσει που έχει διατυπώσει σχετικά η Επιτροπή των Περιφερειών. Η Κομισιόν όμω θεωρεί παρόλα αυτά ότι εξακολουθεί να λειτουργεί καλά το σύστημα. Επιμένετε σε αυτό ή έχετε αλλάξει γνώμη μετά από όλα αυτά. Ο κύριο ε, Φερέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη συζήτηση αυτή για την εφαρμογή της αρχής επικορικότητος τίθεται ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Είναι γεγονός ότι όλη η δυναμική της ε, ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το νομικό πλαίσιο με τη συνδίκη της Αβώνας, αλλά κυρίως η πρακτική εφαρμογή αυτών των αρχών υπονομεύουν σε μεγάλο βαθμό την αρχή της επικορικότητας. Έχουν γυρίσει ανάποδα την έννοια της επικουρικότητα. Γιατί έτσι είναι το κράτος το αποφασίζει ενώ το κράτο ήταν αυτό που έπρεπε να αποφασίζει τι θέλει να κάνει, τώρα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να αποφασίζει τι είναι καλύτερο να το κάνει αυτή. Μπορεί ένα κράτο βέβαια να έχει αντιρρήσει, αλλά το σύστημα ελέγχου δεν δίδει τι απαραίτητε εγγύησει. Οι προποθέσει οι οποίε ε, τίθενται <clears throat> και η όθηση προ μία φεδεραλιστική αντιμετώπιση ουσιαστικά εμποδίσουν τα κράτη-μέλη να αντιδράσουν ακόμα και όταν παραβιάζονται οι αρχές της επικουρικότητας. Γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα επανέλθουμε και πάλι στην αρχή της επικουρικότητας και να σα δώσουμε το πραγματικό της περιεχόμενο, δηλαδή ότι είναι οι λαοί οι οποίοι αποφασίζουν τι πρέπει να γίνεται σε ενωσιακό επίπεδο και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα επιβάλλει στους λαούς αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι το καλύτερο να γίνει για αυτός και το συμφέρον τους. Ευχαριστώ. Κύριο Στογιάννοφ για ένα λεπτό. Monsieur Έχετε το λόγο κυρία Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω πως ε, η αρχή σύμφωνα με την οποία τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να επικαλεστούν την αρχή της επικουρικότητας δεν λειτουργεί σωστά. Δύο χρόνια μετά τη θέση ενισχύ της ε, συνθήκης Λισαβόνας τα εθνικά κοινοβούλια ποτέ δεν έχουν φέρει κάποια αντίρρηση σε βαθμό επαρκή για να σταματήσει η εφαρμογή αυτής της αρχής και μάλιστα αυτό είχε συμπεριληφθεί στη συνθήκη της Λισαβόνας γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι δεν θα λειτουργούσε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πως η κοινοβουλευτική διαδικασία χρειάζεται χρόνο και μιλάμε μόνο για ένα κοινοβούλιο. Οπότε φαντάζεστε τι θα γίνει με 27 κοινοβούλια. Οπότε θεωρώ πως η αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι ε, η εξή πρώτα απ' όλα να έχουμε την έγκριση των Εθνικών Κοινοβουλίων και μετά να εγκρίνουμε το νόμο. Σας ευχαριστώ κύριο Σκέλη, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, η αρχή της ε, επικουρικότητας είναι μάλλον μία από τις αρχές οποίες επικαλούμαστε πιο συχνά. Είναι επίσης δύναμη και αδυναμία. Είναι δύναμη υπό την έννοια πως τα κράτη-μέλη μπορούν να νομοθετήσουν ε, σε κάποιους τομείς από μόνοι τους και δεν χρειάζεται να φορτώνουν τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αδυναμία και είναι αδυναμία όπως βλέπουμε ε, την απάντηση στην οικονομική κρίση, καθώς τα πράγματα θα έπρεπε να γίνουν πολύ πιο γρήγορα, αλλά λόγω της επικουρικότητας αυτό δεν γίνεται. Όμως, εάν προχωρήσουμε σε αλλαγή της συνθήκης, θα πρέπει να ορίσουμε επακριβώς και να προσέξουμε πάρα πολύ και να συνεργαστούμε με τα εθνικά κοινοβούλια για να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Του τουλεχθέντο είναι ενθαρρυντικό να ακούμε αυτά τα οποία είπε ο κύριο Επίτροπο όσον αφορά τι απαντήσει από τα εθνικά κοινοβούλια σε σχέση με τη συνθήκη τη Λισαβόνα και την επικουρικότητα και αυτή είναι η εμπειρία μου και από τη δική μου χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σεύκοβιτς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου για τις απαντήσεις τους και για τις εισαγωγικές τους ε, παρατηρήσεις και να ευχαριστήσω και όλο το σύνολο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επικοδομητική του προσέγγιση σε αυτό το μηχανισμό και για τη συνεργασία που έχει δώσει στα Εθνικά Κοινοβούλια και στην Κομισιόν στο πλαίσιο αυτό, γιατί είμαι πεπισμένος ότι ε, μπορεί να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά ο μηχανισμός ελέγχου της επικουρικότητας προς το συμφέρον όλων μας. Αυτό δεν είναι για να μπλοκάρουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά για να την κάνουμε πιο διάφανη στους πολίτες και πιο δημοκρατική διότι τα θέματα αυτά με τον τρόπο αυτό μπορούν να έρθουν κοντύτερα στους πολίτες και στις καρδιές τους. Και πρέπει να τονίσω ότι χαιρετίζω ιδιαίτερα το θετικό τόνο και την επικοδομητική προσέγγιση που έχουν ακολουθήσει οι ομιλητές, οι, συγγνώμη, οι επικεφαλής των Εθνικών Κοινοβουλίων σε όλο αυτό το θέμα, γιατί αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να έχουμε μια περιεκτική Ευρώπη η οποία είναι πράγματι συνδεδεμένη και με τις ανησυχίες και τους πόθους των πολιτών μας. Η Κομισιόν βρίσκεται σε ενεργό πολιτικό διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια, ο οποίο ήταν ιδιαίτερα καρποφόρος, όπως προσπάθησε να δείξω και με τον αριθμό των ε, αιτιολογημένων γνωμών και γνωμοδοτήσεων που δόθηκαν. Ελπίζουμε θα συνεχίσει αυτή η διαδικασία και στο μέλλον. Το, μέλλον, το ερώτημα τώρα που έχει να κάνει με την ε, αντιμετώπιση της Επιτροπής Περιφερειών. Προφανώς συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την Επιτροπή των Περιφερειών η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στο να ακούγεται η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο ειδικά η Επιτροπή των Περιφερειών έχει ένα δίκτυο εποπτείας της επικουρικότητας που είναι το σημείο επαφή για τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ και δίνει τη δυνατότητα στην Κομισιόν σε ορισμένε περιπτώσει να ενισχύσει την ανάλυση και ανατομή των περιφερειακών πτυχών των νομοθετημάτων του. Επίση, βοηθάει την Κομισιόν να αναλύσει την εφαρμογή τη αρχή τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα και το πράττει και στο μέλλον. Πρέπει να πω ότι βάσει βάση του πρωτοκόλου συνεργασία μεταξύ τη Επιτροπή και τη Επιτροπή των Περιφερειών, η Κομισιόν δίδει τακτικά στην Επιτροπή Περιφερειών τα σχόλιά τη σε σχέση με τι γνωμοδοτήσει σε ό,τι αφορά τώρα τον έλεγχο της επικουρικότητας και τον μηχανισμό ελέγχου από τα Εθνικά Κοινοβούλια και τη συμμετοχή των περιφερειακών νομοθετικών σωμάτων, θα πρέπει να σεβαστούμε τη συνθήκη. Η συνθήκη είναι πάρα πολύ σαφής και επακριβής. Λέει ότι κάθε εθνικό κοινοβούλιο <clears throat> έχει τη δυνατότητα και την διακριτική ευχέρεια να ζητά τη διαβούλευση με περιφερειακά κοινοβούλια και πρέπει να σεβαστούμε λοιπόν αυτή την ρήτρα των συνθήκων. Πώ λειτουργεί τώρα αυτό ο μηχανισμό στην πράξη. Αυτό ήταν το πρώτο και το τελευταίο ερώτημα που ετέθη. Πρέπει να σα πω ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν σταθεί πάρα πολύ αποτελεσματικά στο να δώσουν μια απάντηση στις νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν. Δεν φαίνεται να έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με το να σέβονται την προθεσμία των 8 εβδομάδων και δεν χρειάζεται να φτάσουν στα όρια αυτών των προθεσμιών. Όταν στέλνετε μια πρόταση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, στέλνετε, αποστέλλετε και στα Εθνικά Κοινοβούλια και μέσα σε 8 εβδομάδες τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι έτοιμα να μας δώσουν τις απόψεις τους για τα θέματα αυτά. Αυτό το οποίο προσπαθούμε τώρα να επιτύχουμε από την πλευρά της Κομισιόν είναι να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στις απαντήσεις μας. Έχουμε ένα νέο μηχανογραφικό σύστημα το οποίο κάνει καλύτερη καταγραφή όλων των απαντήσεων και προσπαθούμε να βελτιώσουμε και την ποιότητα των απαντήσεών μας προς τα Εθνικά Κοινοβούλια και να εξασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο εποφελώς τις απαντήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων. Νομίζω λοιπόν ότι μετά την θέση εφαρμογής τη συνθήκη Λισαβόνα δουλεύει μια χαρά ο μηχανισμό ελέγχου τη επικουρικότητα και θα είναι και στο μέλλον ένα σημαντικό τρόπο για να πλησιάσουν τα εθνικά κοινοβούλια στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Κλείνει και αυτή η συζήτηση. Η επόμενη συνεδρία σε ολομέλεια είναι αύριο στι 9 η ώρα μέχρι τις 1.30 η μέση διάταξη έχει δημοσιευτεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Τέλος της συνεδρίασης. Καλό βράδυ σε όλους.